catch this, the eye ή των παρεμβάσεων ενός λεπτού θα πρέπει να διακόψω τη συνεδρίαση έως η κυρία Κορνέλισον όμω ήρθε, οπότε θα πρεπει να διακοψω τη συνεδριαση εως η κυρια Κορνέλη κορνελισον όμως ηρθε οποτε θα δουμε τι γίνεται με τη δική της έκθεση, παρουσίαση των δικαιωμάτων των γενικών σε 56 Παλαιστινίες Παρακαλώ, καθίστε και έχετε το λόγο. Κυρία Κονέλη, σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά. Και μόλις ε, έρχομαι από ψηφοφορία και με συγχωρείτε για την ε, καθυστέρηση. Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάστηκαν μαζί μου. Υπάρχουν βεβαίως οι σκιώδεις η γραμματεία της Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σε κάθε φάση αυτής της ε, έκθεσης ε, μας ε, συμβούλευε και πραγματικά ήταν εξαιρετικό το έργο της. Επίσης όλες οι κυβερνήσεις των Βαλκανικών κρατών αντέδρασαν Πολλές ΜΚΟ επίσης, τουλάχιστον 24, ε, υπηρεσίες διάφορες, ε, πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν. Υπ' αυτή την έννοια, ακόμα και πριν την ε, ψηφοφορία, ήδη η έκθεση αυτή έχει επιτύχει το στόχο της, γιατί είχαμε μια ευρύτατη συζήτηση για τα δικαιώματα των γυναικών και ήδη Βλέπω πως έχει υιοθετηθεί. Οι ΜΚΟ χρησιμοποιούν την έκθεση για τους στόχους τους. Με έχουν ήδη προσκαλέσει σε κάποια κοινοβούλια για να μιλήσω για την έκθεση μετά την ευριανή ψηφοφορία και χαίρομαι για το ότι μπορώ να πω πως ήδη μεταξύ του σχεδίου και της έκθεσης η οποία θα ψηφιστεί τελικά μπορέσαμε να σβήσουμε κάποιες συστάσεις για την Κροατία γιατί έκαναν αυτά τα οποία ε, συστήναμε. Και θα ήθελα τα επόμενα χρόνια να φύγουν όλες οι συστάσεις γιατί όλες οι χώρες πραγματικά προσπαθούν να προωθήσουν τα δικαιώματα των γυναικών. Το σημαντικότερο θέμα εδώ πέρα είναι πως πολλά τέτοια δικαιώματα υπάρχουν τώρα στα χαρτιά. Οι χώρες των Βαλκανίων ε, προσπαθούν να υιοθετήσουν νομοθεσία που θα είναι σύμφωνη με το κοινοτικό κεκτημένο. Στην πράξη όμως ε, δεν ε, μπορούν να τα εκμεταλλευτούν αυτά τα δικαιώματα, να τα ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα οι γυναίκες, είτε γιατί δεν το γνωρίζουν, είτε γιατί δεν ξέρουν πού μπορούν να καταγγείλουν τη διακριτική μεταχείριση, είτε γιατί το κράτος δικαίου δεν λειτουργεί ως όφιλε για τις γυναίκες. Με τις συστάσεις μας αυτές λοιπόν δεν κάναμε κάποιες γενικές στάσεις για όλες τις χώρες αλλά κάναμε και συγκεκριμένες αναχώρα των Δυτικών Βαλκανίων. Ελπίζω λοιπόν να ανταποκριθούν και να αρχίσουν να τις εφαρμόζουν. Κάτι άλλο. που υποσχέθηκα στους συναδέλφους. Ε, είχαμε μια συζήτηση για το πώς θα αποκαλέσουμε μια χώρα. Αν θα ήταν η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ή να αφήσουμε το ε, πρώτο μέρος, το πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία. Τελικά καταλήξαμε σε ένα συμβιβασμό και αποφασίσαμε το ουσιαστικό να είναι η Πουγουδουμού και το επίθετο να είναι ο Μακεδόνας ή Μακεδονικός. Ελπίζω λοιπόν να είναι όλοι ικανοποιημένοι σε, όλες, σε όλα τα κρατημέλη αλλά και στην λόγω χώρα. Μου επισήμαναν πως ε, δεν γίνεται αυτό σε όλες τις γλώσσες. Ε, ελπίζω να λυθεί και αυτό το πρόβλημα και να είναι όλοι ικανοποιημένοι και να υπερψηφίσουν την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νίλσεν. Τώρα περνάμε αμέσως στο θέμα, στη διαδικασία του ΚΑΤΣΤΙΑΙ και θα δώσω το λόγο στην κυρία Σεπιντέσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ω προ την έκθεση αυτή, θα ήθελα να παρουσιάσω τη θέση μα για το θέμα τη ανισότητα ε, μεταχείριση των γυναικών στι χώρε των ε, Δυτικών Βαλκανίων. Νομίζω ότι πρόκειται για κάτι που έχει πολιτιστικά αίτια, όμως άντρες και γυναίκες που τόσο πολύ ενεργοποιούνται στην αγορά εργασίας, σε μια ελεύθερη αγορά θα πρέπει να καταπολεμήσουν τα στερεότυπα κατά των γυναικών. Διότι η κοινωνική ε, καθιέρωση αυτής της άνησης μεταχείρισης σε κοινωνικό επίπεδο είναι κάτι που πραγματικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ακόμη και κάποια περιστατικά βία καταγράφονται κατά των γυναικών. Πράγματα που σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορεί να γίνουν ανεκτά. Θα πρέπει να ζητηθεί από τι κυβερνήσει των χωρών αυτών να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την άνηση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Γιατί θα πρέπει να δοθεί κάποια απόκριση για τι περιπτώσει αυτέ και να μπορέσουμε και εμεί να συμβάλλουμε στην πληθύνση τη θέση των γυναικών στι χώρε αυτέ. Ευχαριστούμε, κυρία Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, δεν υπάρχουν αρκετά στατιστικά στοιχεία για την ισότητα μεταξύ των φίλων, τη βία κατά των γυναικών την παραβίαση των δικαιωμάτων τους ε, στις χώρες ε, βαλκανικές ε, που υποψήφιες για ένταξη. Χρειαζόμαστε όμως αυτά τα στοιχεία για να βελτιώσουμε τις συνθήκες των γυναικών που είναι θύματα πολλαπλών διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να παρακολουθήσει το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών και να ενημερώνει για τη βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων. Πρέπει επίσης να προωθήσουμε τη συμμετοχή του στην αγορά εργασίας και μια ισότιμη ε, συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Επίσης πρέπει να προωθήσουμε το επιχειρηματικό πνεύμα στις γυναίκες που είναι σημαντικό για την ε, ανάπτυξη, για την ενίσχυση της δημοκρατίας στις χώρες που υποψήφιες για ένταξη. Ευχαριστώ κυρία Βέρτμαν. ευχαριστώ. Πάρα πολλοί άνθρωποι εργάζονται πάρα πολύ σκληρά για... και εμείς εργαστήκαμε σκληρά για να εγκρίνουμε τις ε, διατάξεις αυτές για την προστασία των γυναικών. Όμως ε, πετούνται κάποια βήματα ακόμα. Οι χώρες αυτές, όπως είπαμε, βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία όσον αφορά την πρόοδό τους και Βεβαίω θα ήθελα συνολικά να πω στου αδέλφου πω πρόκειται για μια αντικειμενική, ισορροπημένη ε, έκθεση και με ικανοποίησε ε, ιδιαίτερα το ότι σημειώνεται η πρόοδο η οποία έχει σημειωθεί. Γι' αυτό το θέμα ότι τις χώρε αυτέ να εντείνουν τις ε, προσπάθειε του Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, την εισηγητρία και για την εξαιρετική ε, έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντικό να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, στον ρόλο των γυναικών και στα Δυτικά Βαλκάνια και οπουδήποτε αλλού άλλωστε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά από τους πολέμους της δεκαετίας του 90 να ε, εστιάσουμε στην ε, δυνατότητα στην, στις γυναίκες και τη συμμετοχή τους ε, στα κοινοβούλια άσχετα από την ε, ηθαγένειά τους οι εγκληματίες πολέμου δεν έχουν ε, τιμωρηθεί υπάρχουν γυναίκες που έχουν βιαστεί στη διάρκεια των πολέμων Άρα η πολιτική συμμετοχή των γυναικών είναι πάρα πολύ σημαντική. Στο κοσυφοπαίδιο ε, υπάρχει ένα τρίτο των γυναικών, των βουλευτών που είναι ε, γυναίκες και αυτό πρέπει να γίνει και στις άλλες χώρες. Ο κύριος Πασκά. Ευχαριστώ πολύ Καταλαβαίνω την προσέγγιση της κυρίας κονέλησεν σχετικά με τις γυναίκες και το σεβασμό των δικαιωμάτων τους στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις διαφορές μεταξύ της έκθεσης αυτής και το, ε, της έκθεσης ε, του περασμένου μήνα ζητήσαμε από το Κοινοβούλιο του Κοσφοπεδίου του Κόσοβο να είναι πιο ενεργό, να καταβάλουν προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν ορισμένα προβλήματα όπως το εμπόριο ανθρώπων αν θέλετε και μιλήσαμε και για το ότι πρέπει να εκπροσωπούνται πολύ περισσότερο οι γυναίκες σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Είναι λοιπόν πολύ παρακολουθή να υπάρχουν διαφορές. Θα έπρεπε να είναι ίδιες οι εκθέσεις για το ίδιο θέμα. Το κάνουν. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Η παραδοσιακή προσέγγιση που υπάρχει στα Δυτικά Βαλκάνια για το ρόλο της γυναίκας είναι τέτοια που ε, χρειάζεται βελτίωση και εξυγχρονισμό για να γίνουν οι χώρες αυτές μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει τέτοιες προσπάθειες. Όμως αναρωτιέμαι κατά πόσον θα πρέπει αυτό να γίνει με θετική θετική με θετικές διακρίσεις και ποσοστός για τις γυναίκες ή με άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες θα καταργήσουν την άνηση μεταχείριση και τα κλισέ που υπάρχουν στις χώρες αυτές. Παραδείγματος χάνει ενίσχυση επιχειρηματικότητας των γυναικών. Ε, η ίσως ε, θα πρέπει επίσης να πούμε γιατί ήρθαμε σε επαφή με εκπροσώπους από πολλές χώρες ε, ότι θα χαιρετίζαν τις πρωτοβουλίες αυτές και ίσως δεν θέλουν θετικές διακρίσεις και ποσοστώσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για μια πολύ καλή έκθεση η οποία δίνει έμφαση στην ισότητα και στο νόημα της ε, ισότητας και των δικαιωμάτων των γυναικών στις χώρες προσχώρησης από τα Βαλκάνια. Βελτιώνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα στις χώρες των Βαλκανίων. από τις μείζονες προκλήσεις εξακολουθεί ο αριθμός των γυναικών στην αγορά εργασίας που είναι μικρός. Εξαρτώνται δηλαδή οικονομικά πολλές γυναίκες από τους άνδρες. Επίσης και σε θέσεις ε, σημαντικές για λήψη αποφάσεων ή στην οικονομία οι γυναίκες είναι λίγες. Για να έχουμε λοιπόν ισότητα στους τομείς αυτούς θα πρέπει να υλοποιήσουμε τις ποσοστώσεις. Ήδη μια χώρα το έχει πράξει, άλλες όχι όμως. Θα πρέπει τα στερεότυπα επίσης να καταργηθούν στι χώρες αυτές. Είναι καιρό για τις κυβερνήσεις των κρατών αυτών να δεσμευτούν ότι θα σέβονται τα διεθνή πρότυπα, όχι μόνο στην πολιτική αλλά και στην οικονομία. Όπως είπε η συγγήτρια, άλλο είναι η θεωρία, άλλο είναι η πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λούαν. Κυρία Πρόεδρε, το θέμα της ισότητας στις υποψήφιες χώρες δεν είναι κάτι που ταιριάζει σε θέση με τις παρούσες χώρες μέλη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή σε αυτές τις χώρες είναι κάτι απαραίτητο για σταθεροποίηση της κατάστασης και την ομαλοποίηση την εξομάλυνση σε αυτές τις χώρες και να επιταχύνει την προσχώρησή τους. Είναι απαράδεκτο ότι μέχρι τώρα, κυρίως στην Ήπεθρο, Πολλές γυναίκες εξακολουθούν να είναι θύματα διάκρισης για λόγους θρησκευτικού, για λόγους εθνοτικούς. Λείπουν νομικά μέσα για την καταπολέμηση του φαινομένου και την καταπολέμηση της οικιακής βίας. Η έλλειψη της αντισύλληψης επίσης είναι άλλο στοιχείο που δυσκολεύει τη ζωή των γυναικών και δεν γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Θα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματική βαθμολόγηση των χωρών αυτών και να γίνει και νομική μεταρρύθμιση με στόχο την εφαρμογή των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ισότητα των φίλων, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λούαν. Ο κύριος Κονφεράτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το θέμα των δικαιωμάτων γυναικών είναι πάντα σημαντικό θέμα και τώρα περισσότερο όσον αφορά μάλιστα χώρες οι οποίες βρίσκονται στα πρόθυρα της ε, εξομάλυνσης και της εδραίωσης της δημοκρατίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα να παρατηρηθεί και όσον αφορά το θέμα της ηθαγένειας και στο επίπεδο όμως του χώρου εργασίας. Αντικειμενικά είναι αδύναμες οι γυναίκες, αδύναμες θέσει στον τόπο εργασίας, ακόμα περισσότερο όταν έχουν και βία, αντιμετωπίζουν βία στις, στα σπίτια τους. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο φαινόμενο όσα αφορούν τις λεπτομέρειες και το περιεχόμενο της εργατικής δραστηριότητα των γυναικών. Πολύ συχνά έχουν πρόβλημα να βρουν δουλειά. Και είναι μια δουλειά φτωχή πολύ συχνά, διότι δεν έχουν επαρκής γνώση αυτές οι γυναίκες. Και είναι σε ακόμα δυσχερέστερη θέση οι γυναίκες όταν δουλεύουν, είναι αντικείμενο διάκρισης σχέση με τους άντρες όσον αφορά την αμοιβή και τα δικαιώματα. Είναι ευκταίο να εξετάσουμε το θέμα της ε, ηθαγένεια και των δικαιωμάτων που έχουν οι γυναίκες και ταυτόχρονα με το, τα δικαιώματα που έχουν στο χώρο εργασίας. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστούμε την συγγήτρια για την πολύ καλή δουλειά που έκανε στο θέμα. Η ισότητα είναι κάτι που ενστεριζόμαστε όλοι. Δυστυχώς όμως δεν εφαρμόζεται η ισότητα στην πράξη. Ε, κυρίως αν δει, τι γίνεται εδώ την πέμπτη, το πέμπτη απόγευμα που ασχολούμαστε με ανθρώπινα δικαιώματα και βλέπουμε ότι σε κάποιες χώρες έχουν ελάχιστα δικαιώματα γυναίκες. Προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Και εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχουμε ισότητα επισήμω. Οι δυνατότητε όμω για τι γυναίκε να προοδεύσουν είναι πολύ λίγε. Υπάρχουν ε, φραγμοί που συζητήσαμε Δυνατότητε για να κινηθούν στον πολιτικό κόσμο και λοιπά και στα διοικητικά συμβούλια. Γι' αυτό θα πρέπει οι χώρες υποψήφιες προσχώρηση να έχουν προτεραιότητα την ισότητα και θα πρέπει να σημειώσουν πρόοδο σε αυτόν τον τομέα για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι θα πρέπει να τους πούμε ότι δεν θα τους επιτρέψουμε να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπω τον κύριο Πόρες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική της δουλειά. Όποτε μιλούμε για δικαιώματα των γυναικών, θα πρέπει να θυμόμαστε και την ιστορία των Βαλκανίων. Εν μέρη, ε, είναι, κάποιες μάλλον από τις χώρες είναι μέλη της Ένωσης, κάποιες είναι υποψήφιες για ένταξη. Έχουν ένα παρελθόν ε, δύσκολο με το οποίο πρέπει να συμβιλωθούν οι χώρες αυτές. Ε, ε, στο μεταπολεμικό αυτό στάδιο και σε ό,τι αφορά τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών. Όμω τώρα πρέπει να ανταλλάσσουμε πλέον καλέ πρακτικέ, εμπειρίε και είναι καιρό να προωθήσουμε και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών και στο δημόσιο βίο. Επίσης να προωθήσουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στα ανώτερα κλιμάκια τη διοίκηση. Τι καλέ πρακτικέ τι έχουμε, τι βέλτιστε πρακτικέ. Πρέπει απλά να τι προωθήσουμε πρέπει να προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε όλα τα κράτη των Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικές για τα δύο φύλλα, ενσωμάτωση της διάστασης του φίλου είναι σημαντικές ε, συνιστώσεις και εμείς πρέπει να δώσουμε ε, το καλό παράδειγμα όταν εκπονούμε ε, τη σχετική νομοθεσία ώστε να μπορέσουμε να τους ζητάμε μετά να προσαρμόσουν την νομοθεσία τους στη δική μας. <clears throat> Thank you all. Now, this is... Σας ευχαριστώ πολύ. Επίτροπος ε, Κρούς τώρα. Thank you, President. Honorable members. Τα δύσκολα σε εσάς, κυρία Κρούς. Κυρία Κρούς, Καλώς ορίζω και εγώ την ε, έκθεση της κυρίας Κορνέλισεν για τα δικαιώματα των γενικών συμπορέντας και βαλκανικές χώρες. Χαίρομαι γιατί λαμβάνετε υπόψη σας ε, πολλούς εμπλεκομένους φορείς, οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών, βουλευτές, προσώπους των κυβερνήσεων, μεταξύ άλλων και στην έκθεσή σας εντοπίζετε ζητήματα που και η Κομισιόν θεωρεί σημαντικά για την αξιολόγηση της πρόοδου που γίνεται σε αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων. Όπω αναφέρει κύριε Πρόεδρε και η έκθεση, η υλοποίηση, η επιβολή τη νομοθεσία ε, στον τομέα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώ για αυτό το λόγο και βοηθά στη μεταφορά του κεκτημένου για την ισότητα των φύλων στο εθνικό δίκαιο των υποψηφίων και δυνητικά υποψηφίων χωρών, αλλά παρέχει επίση και οικονομική υποστήριξη και ελέγχει, παρακολουθεί την εφαρμογή και την επιβολή της εθνικής νομοθεσίας μέσω των διαφόρων μέσων της προταξιακή στρατηγικής. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η πλήρης μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η επιβολή όλων των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ισότητας των δύο φύλων είναι και αυστηρή προϋπόθεση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζωτική σημασία επίσης είναι η ανάπτυξη των θεσμικών και διοικητικών δομών που θα διευκολύνουν την εφαρμογή και την επιβολή των δικαιωμάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνει την εστίαση, την μεγαλύτερη εστίαση στην ισότητα των δυοφύλων και στα δικαιώματα των γυναικών στι χώρε των Βαλκανίων. Για παράδειγμα, παράσχα ε, βοήθεια για την εκπαίδευση των δικαστών και συνεργαζόμαστε και με πολλέ οργανώσει που ασχολούνται με την ισότητα των δύο Το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μπορεί να ε, δώσει άμεσα χρηματοδότηση σε γυναικές οργανώσεις και έχουν ωφεληθεί τα μάλα οι οργανώσεις αυτές. Επίσης, οι ε, πρωτοβουλίες ε, που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα, προωθούνται. Ενισχύονται, χρηματοδοτούνται προγράμματα στον τομέα αυτό. Το 2011 είχαμε ήδη προτείνει μια καινοτόμο προσέγγιση για του τομεί ε, τη δικαιοσύνη και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η στρατηγική αυτή είχε παρουσιάσει και έναν πιο ισχυρό μηχανισμό. Και το κεφάλαιο 24 για τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια και το κεφάλαιο 23 για τα δικαστικό σώμα και τα θεμελιώδη δικαιώματα έγιναν σημαντικά κίνητρα προς μεταρρύθμιση. Το κεφάλαιο 23 είναι μεταξύ των πρώτων που ανοίγει και μεταξύ των τελευταίων που κλείνει. Πρώτα πρέπει να επιβεβαιωθεί ε, ότι υπάρχουν απαραίτητε μεταρρυθμίσει και πρόοδο στον τομέα. Ολοκληρώνοντα, θέλω να πω ότι με, με ικανοποίηση σημειώνουμε ότι η Κροατία, μελλοντικό μέλο τη Ένωση, πλήρω ε, ευθυγραμμίστηκε ε, με την ομοθεσία στον τομέα της των δύο φύλων. Και αυτό που είπατε μπορώ να το καλωσορίσω θερμά. Δηλαδή θα μπορούσε η Κροατία να αποτελέσει ένα παράδειγμα για ολόκληρη την περιοχή. Είναι ένα ακόμη παράδειγμα της ε, ε, μεταμορφωτικής δύναμης που έχει η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συναδέλφους, ιδιαίτερα την εισηγήτρια. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12.30. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε στην έκθεση της κυρίας Βέιμπερ για το χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρυθμίσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Βέμπερ,